Περνάω στο επόμενο θέμα. Η υπογραφή πράξεων σύμφωνα με την κανονική νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 74 το περιεχόμενο θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής και θα το ελέγξετε. Πήρα επίσης πληροφορίες από την ομάδα των Πασίνων την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ότι ο κύριος Φίλιπ Λάμπερτς αντικαθιστά την Εύα Ζολή στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση πάνω στην ανακοίνωση της ομάδας των Πρασίνων. Όχι. Αλλαγές τώρα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίες και κύριοι, Θα ξεκινήσω από τη Δευτέρα. Η ομάδα των φιλελευθέρων, όχι διορθώνω, η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ζήτησε η έκθεση Γκάλο να μην τεθεί προς Αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Ο κύριος Σούλτσο θέτει το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η κοινοβουλευτική μας ομάδα ήδη στην διάσκεψη των Προέδρων την προηγούμενη εβδομάδα επεσήμανε ότι η έκθεση Γκαλό είναι πολύ επίμαχη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας στο Σώμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την περαιτέρω εξέταση αυτής της έκθεσης, θα έπρεπε για άλλη μία φορά να εξεταθεί σε βάθος